Varmt välkomna till dagens utskottsmöte med jämställdhetsutskottet. Καλημέρα σας, σας καλωσορίζω σε αυτή τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας για τις ίσες ευκαιρίες. Καλωσορίζω και τους υπαλλήλους και τους επισκέπτες. Καλωσορίζω επίσης και τους διερμηνείς διότι χάρη σε αυτούς και αυτές καταλαβαίνόμαστε. Για να δούμε τι λέει η μερίσια διάταξη. Σημειώστε παρακαλώ ότι η ψηφοφορία της έκθεσης της κυρίας Κώστας για το οργανωμένο έγκλημα, το σημείο 12 δηλαδή, θα γίνει αμέσως μετά το 8 σημειώστε το παρακαλώ το 12 αμέσως μετά το 8 και με την τροποποίηση αυτή εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Μάλιστα, το 2 τώρα, ανακοινώσει της Προέδρου. Μία ανακοίνωση έχω και εδώ παρακαλώ να σημειώσετε. Προβλέπουμε κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Ανάπτυξης στις 11 σήμερα. Το θέμα είναι η σεξουαλική βία σε πλαίσιο ένοπλης σύραξη. ιδιαίτερα δεν στο Κονγκό, στο Δημοκρατία του Κονγκό. Κοινή λοιπόν συνεδρίαση με την Επιτροπή Ανάπτυξης θα έρθει εκεί η ειδική εκπρόσωπος του ΟΗΕ για την καταπολέμηση το, της σεξουαλικής βίας σε περίπτωση ένοπλης σύραξης και θα αλλάξουμε αίθουσα, θα φύγουμε από εδώ και θα πάμε στην αίθουσα 3Z2 του κτηρίου ΑΣΠ. 3Z2 στις 11. Ελπίζω να έρθετε πολύ εκεί, στην κοινή αυτή συνεδρίαση. Στις 11 επαναλαμβάνω. Αυτό είχα να σας πω. Περνούμε στο 3. Πρόκειται για την απόφαση του δικαστηρίου στην υπόθεση σε 236 κάθετος 09. Βελγική Ένωση Καταναλωτών Τέστασα κατά Συμβουλίου Υπουργών. Το κριτήριο του φύλου ως συντελεστής αξιολόγησης των ασφαλιστικών κινδύνων. Θα γίνει λοιπόν μια ανταλλαγή απόψεων για αυτό το θέμα σήμερα και θα πρόκειται για ένα πρώτο βήμα της επεξεργασίας από μας μιας έκθεσης πρωτοβουλίας που θα αφορά ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο η απόφαση αυτή και η σχετική οδηγία θα εφαρμοστούν. Γιατί η Επιτροπή μας αποφάσισε να κάνει αυτή, την ασυγράψη, αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας. Η κυρία Ντουρμάη την έχει αναλάβει. Ξέρουμε ότι η Κομισιόν επίσης προετοιμάζει μια μελέτη, μια έκθεση για τον τρόπο εφαρμογής της σχετικής οδηγίας και θα γίνει και αυτό μέσα στο χρόνο. Στα πλαίσια λοιπόν της εφαρμογής της οδηγίας πρέπει να λάβουμε υπόψη και αυτή την απόφαση του δικαστηρίου. Σας είχα πει τον αριθμό προηγουμένως. Δυστυχώς ε, οι εκπρόσωποι του τεστ δεν μπόρεσαν να προσέλθουν σήμερα. Είχαν έρθει άλλη φορά προηγούμενη, αλλά σήμερα δεν μπόρεσαν. Θα ακούσουμε όμως εκπρόσωπο της Κομισιόν και επίσης εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασφαλιστών και Επανασφαλιστών. και θα αρχίσουμε τη συζήτηση ακούγοντας τους δύο αυτούς εκπροσώπους. Και μετά θα ακούσουμε και την εισηγήτριά μας την κυρία Ντορμάη και θα αρχίσει η συζήτηση. Πρώτα πρώτα λοιπόν η Κομισιόν. κυρία Κριστίν Τομπόη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, χαίρομαι που μπορώ να συμμετάσχω στη συζήτηση για αυτή την πολύ σημαντική απόφαση ε, διότι δεν θα μακρηγορήσω επειδή πρέπει να έχουμε μία συζήτηση μεταξύ μας. Θέλω πλούστατα να σας πω ποια είναι τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά και ε, τι συμπεράσματα αποκομίζουμε και επίσης να σας δώσω μία ιδέα σχετικά με τα επόμενα βήματα τα οποία πρόκειται να αναλυθούν από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ουσιαστικά αναφερόμαστε στο γεγονός ότι πρόκειται για την οδηγία του 2004 σχετικά με την πρόσβαση σε ε, ε, αγαθά και υπηρεσίες και αυτό αναφέρεται και στον οικονομικό, το χρηματοοικονομικό τομέα και στις ασφάλειες και ιδίως το άρθρο 5 αναφέρεται στην ασφάλιση και περιλαμβάνει δύο ουσιαστικές διατάξεις και θα αναφερθώ πρώτα σε αυτές τις δύο με τις οποίες ασχολούμεθα εδώ. Καταρχήν στο άρθρο 5.1 της βασικές αρχές ε, που είναι ε, ένας κανόνας unisex όπου η ισότητα των φύλων δεν πρέπει να οδηγεί σε ένα διαχωρισμό ε, λόγω του φύλου όσον αφορά τα ασφάλιστρα. Αυτό είναι η βασική αρχή. Και το δεύτερο στοιχείο, το άρθρο 5.2, είναι ε, μία απόκληση από αυτόν τον κανόνα που επιτρέπει υπό συγκεκριμένε προϋποθέσεις να υπάρξει μία διαφοροποίηση μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ε, θέλω να σας πω ότι ουσιαστικά κατά αυτόν τον ε, τρόπο δεν εμποδίζεται να χρησιμοποιηθεί αυτός ο παράγοντας, απλούστατα δεν πρέπει να οδηγεί σε διαφοροποίηση των ασφαλίστρων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και η παρέκκληση του άρθρου 2 ουσιαστικά ε, κηρύχθηκε ε, άκυρη από το δικαστήριο από το 2012. Και για να υπογράψω, για να υπογραμμίσω αυτό το βασικό θέμα και την απόφαση θα τη συγκρίνω με την γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα ο οποίος ε, είχε εκδώσει την γνωμοδότηση του το Σεπτέμβριο πριν λίγους μήνες και ο οποίος έλεγε ότι ε, η υπάρχει μία ανάλυση ε, ε, ε, των ασφαλιστικών πρακτικών η οποία αξιολόγησε αυτές τις πρακτικές και κατέληξε στο ότι μέχρι ενός σημείου Πρόκειται και πάλι για ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών. Θα επανέλθω στο θέμα αυτό γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπρεπε να υιοθετήσει μία έκθεση μέχρι το τέλος του παρελθόντος έτους και να εστιαστεί στον τομέα των ασφαλίσεων. Οπότε το στοιχείο αυτό δεν θα είναι το μοναδικό στην έκθεση αυτή αλλά θα αποτελέσει ένα βασικό θέμα της εκθέσεως και όταν θα δούμε την γνωμοδότηση θα δούμε ότι ήταν σοφό να περιμένουμε την ε, απόφαση ε, και ε, ότι Γι' αυτό αναφερόμαστε και αξιολογούμε τη δικαστική απόφαση στην έκθεση και καθυστερήσαμε την έκδοση της εκθέσεως. Ε, η ε, ε, απόφαση λοιπόν του δικαστηρίου εξεδόθη το Μάρτιο και στην ουσία διαφέρει κατά τη γνώμη μας από την γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα διότι δεν αναλύει σε εις βάθος κάποιον τομέα και το πώς λειτουργεί τις πρακτικές και ούτω καθεξής για μας είναι μία απόφαση που αναφέρεται στην θέληση του νομοθέτη και πώς η οδηγία έχει καταρτιστεί και αν ε, ε, είναι συνεκτική με ε, τα μέσα τα οποία εφαρμόζει. Εάν λοιπόν κοιτάξετε αυτή την παρέκκληση στο άρθρο 5 παράγραφος 2 αναφέρεται στην ε, συνολική θεώρηση και στο στόχο ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο, ο παράγραφο, άρθρο 5 παράγραφος 1 δηλαδή ίση μεταχείριση μεταξύ των φύλων και μετά ε, αναλύει την παρέκκληση στο άρθρο, την εξαίρεση στο άρθρο της παραγράφου 2 5-2 και ε, βλέπουμε εδώ ότι η εξέριξη αυτή ήταν απλώς μια δυνατότητα που είχε προσφερθεί στα κράτη-μέλη. Δεν είχε διατυπωθεί ε, όπως σε άλλα ε, νομοθετήματα όπου λέγεται ότι η μέθοδος αυτή δεν θα θεωρηθεί σαν διάκριση μεταξύ των φύλων. Εδώ απλώς δίνεται μια δυνατότητα στα κράτη-μέλη και λέγεται ότι ορισμένε Προποθέσει προϋποθέσεις μπορούν να εφαρμόσουν την απόφαση αυτή και αν θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτή την απόφαση θα πρέπει να αποφασίσουν μέχρι κάποια ημερομηνία που ήταν μέχρι το Δεκέμβριο του 2007. Δηλαδή η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί η απόφαση αυτή ήταν χρονικά περιορισμένη μέχρι το 2007 και στην περίπτωση αυτή θα έπρεπε να αναθεωρήσουν την απόφαση αυτή και αυτό που είναι επίσης σημαντικό και ενδιαφέρον είναι ότι στα εκτιμώντας της οδηγίες ε, προβλεπόταν ότι όσοι εφαρμόζουν αυτόν τον κανόνα της ε, ε, ισότητας των φύλων, την παράγραφο 5.1, δεν μπορούσαν να υποφεληθούν της εξαιρέσεως στην παράγραφο 5.2. Οπότε ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, διάφορες εξαιρέσεις ε, στα διάφορα μέσα που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή υπάρχει ένα νόμος από τη μία πλευρά και η πρακτική όπως εφαρμόζεται από την άλλη, αλλά στην περίπτωση αυτή ήταν, υπήρχε ρητή εξαίρεση ευθύς εξ αρχής. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η αρχή των, ε, ε, του κανόνα της ισότητας των φύλων, unisex κατά κάποιον τρόπο ε, λέγεται ότι οι άντρες και οι γυναίκες είναι σε συγκρίσιμη κατάσταση όσον αφορά και τα ασφάλιστρα αλλά και τα ωφέλη από αυτή την ασφάλιση. Δεν υπάρχει διάκριση το εάν η κατάσταση είναι συγκρίσιμη ή όχι είναι ένα ουσιαστικό σημείο διότι εάν δεν είναι συγκρίσιμη η κατάσταση δεν μπορεί να προβεί κανεί στη σύγκριση. Ε, εδώ όμως λέει το δικαστήριο ότι ο νομοθέτης όταν κατήρτισε το νόμο θεώρησε ότι οι άνδρες και οι γυναίκες μπορούν να συγκριθούν στο θέμα αυτό και άρα η εξαίρεση δεν είναι ανοιχτή, ήταν ε, μόνο διαθέσιμη για μια μεταβατική περίοδο. Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε ότι μπορούσαμε να αξιολογήσουμε ε, ότι υπήρχε ε, μία νομοθεσία η οποία ήταν βασική και έπρεπε να είναι και συνεκτική. Ε, για να μπορέσει κανείς να βασιστεί και να καταρτήσει την νομοθεσία επί των αρχών αυτών και ίσως θα χρειαστεί να επανέλθουμε στο θέμα αυτό διότι ε, δεν νομίζω ότι επηρεάζει άλλα θέματα. Ε, εδώ μιλάμε για την ε, νομοθεσία η οποία εφαρμόζεται, για την οδηγία η οποία εφαρμόζεται και περιέχει ορισμένα στοιχεία σχετικά με την ασφάλιση και τις αναπηρίες. Θα είμαι όμως σύντομος και ουσιαστικά θα αναφερθώ στα βασικά βήματα κατά τη γνώμη μας. Καταρχήν θεωρούμε ότι ε, ε, ε, η, απόφαση είναι σαφέστατη όσον αφορά την οδηγία αυτή. Δεν αναφέρομαι υποχρεωτικά στις ε, επιπτώσεις για τα κράτη-μέλη, αλλά η οδηγία λέγει, δηλαδή το δικαστήριο θεωρεί ότι από μία ημερομηνία και πέραν η οδηγία δεν εφαρμόζεται, είναι άκυρη και θα μπορούσαμε να, ε, να παρουσιάσουμε ορισμένες ε, διατάξεις οι οποίες θα ίσχυαν για μένα περιορισμένο χρόνο μόνο διότι η απόφαση είναι σαφέστατη αλλά έχει πολλές επιπτώσεις για τα κράτη-μέλη και για τον ασφαλιστικό κλάδο. Και καλό θα ήταν να ξέρετε ότι κανένα κράτος δεν είχε χρησιμοποιήσει αυτή την εξαίρεση και δεν αναφέρουμε εδώ ε, για όλες τις ασφάλειες ε, αλλά ε, όλα τα κράτη χρησιμοποίησαν την εξαίρεση μόνο για τις ασφάλειες ζωής, για προϊόντα δηλαδή σχετικά με, σχετικά με την ασφάλεια ζωής. Θα υπάρχουν λοιπόν επιπτώσεις και θα επηρεαστεί ο τομέας των ασφαλιών. Τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Καταρχήν θέλουμε να συζητήσουμε με αυτούς οι οποίοι πρέπει να εφαρμόσουν τη δικαστική απόφαση και ε, να δούμε ε, αν ε, υπάρχουν διαφορές μεταξύ προϊόντων, μεταξύ εμπλεκομένων παραγόντων γιατί θέλουμε η έκθεση αυτή να είναι πλήρης σχετικά με την κατάσταση. Η πρώτη ημερομηνία είναι 20 Ιουνίου. Οπότε θα υπάρξει μία συζήτηση με όλους τους ενδιαφερομένους. Θα είναι μία γενική συζήτηση ε, υπομορφήν η οποία χρησιμοποιείται από ετών για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιληφθεί ε, πώς ε, η, ο τομέας των ασφαλιών αντιμετωπίζει την ισότητα των φύλων. Η συνάντηση αυτή θα είναι 20 Ιουνίου και θα συζητήσουμε συζητήσουμε τις ε, πρακτικές επιπτώσεις βάσει ενός ερωτηματολογίου και κατόπιν αξιολογήσεως όλων των ε, γλαπτών ε, απαντήσεων που θα έχουμε μετά τη συζήτηση αυτή. Και στη συνέχεια το Σεπτέμβριο η Επίτροπος θα συναντηθεί με τους ηγέτες από τον ασφαλιστικό κλάδο. Όλες οι διαβουλεύσεις αυτές, οι οποίες θα οργανωθούν στους επόμενους μήνες, θα μας επιτρέψουν να ετοιμάσουμε μία έκθεση και ελπίζουμε η έκθεση αυτή να μπορέσει να υιοθετηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου και να συνοδευτεί από κατευθυντήριες γραμμές για τον ασφαλιστικό τομέα για να διευκρινίσει ορισμένα θέματα και εδώ σταματώ. Ευχαριστώ, κύριε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τόμποη για τις ε, πληροφορίες που μας δώσατε και για να μην ε, καθυστερούμε θα δώσω το λόγο στην κυρία Μικαέλα Κόλλαρ η οποία εκπροσωπεί την Ένωση Ευρωπαίων Ασφαλιστών και Δεύτερα Ασφαλιστών. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Επιτροπή σας και την κυρία Γκουρμάη, την εισηγήτρια που μας κάλεσε εδώ, κάλεσε εδώ την Ομοσπονδία των Ευρωπαϊκών, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Εταιριών. Ε, καλύπτουμε γύρω στο 90% των εταιριών στον κλάδο και είναι πολύ σημαντικό το θέμα που συζητείτε σήμερα, γι' αυτό χαιρόμαστε, βρισκόμαστε εδώ. Ο τομέας μας βεβαίως, ε, θα ήθελα να πω ήδη εξ επαρχής, ότι συμμορφούνται απόλυτα με την αρχή και την ίση μεταχείριση των φύλων. βεβαίω, η πρόσφατη απόφαση του δικαστηρίου δεν δημιουργεί για μα. Δεχόμαστε την απόφαση 100% θεωρούμε ότι συμμορφούμεθα με την ε, βασική αρχή αλλά υπάρχουν κάποια ερωτήματα. Πρώτα πρώτα θα θέλαμε να υπάρχει νομική βεβαιότητα. Όπως είπε και η κυρία Τόμπο με μια έννοια η οδηγία είναι σαφή. Η εξαίρεση συνεδρίαση ε, λίγη στις 21 ε, Δεκεμβρίου ε, 2012 και από εκεί και πέρα θα πρέπει βεβαίως να εκδοθούν οι κατευθυντήριες γραμμές για να δούμε πώς θα εφαρμοστεί πέραν αυτής της ημερομηνία η οδηγία. Βεβαίως υπάρχουν φωνές που λένε ότι αντίθετα με την απόφαση του δικαστηρίου ή με αυτά που λέγονται εκεί ε, θα επηρεαστούν και τα συμβόλαια που ισχύουν αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν είναι κάτι που το δεχόμαστε εμείς και η Κομισιόν θεωρεί ότι πρέπει να διευκρινιστεί το θέμα. Θα ήθελα επίσης να σας δώσω δύο-τρεις ακόμη, να παρουσιάσω λόγους για τους οποίους μας ενδιαφέρει η νομική βεβαιότητα. Δείτε, αν στο μέλλον υποβληθούν, ε, γίνουν αντίστοιχε προσφυγές όπως αυτή του Τέστασα ε, στα διάφορα κράτη-μέλη, τα εθνικά δικαστήρια θα πρέπει να αποφανθούν και βεβαίως ε, θα πρέπει να ε, εξασφαλίσουμε ότι οι αποφάσεις των δικαστηρίων αυτές θα είναι σύμμορφες μεταξύ τους και θα βασίζονται και, στη βασική, και στην, στις βασικές νομικές αρχές που ισχύουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Εκείνο το οποίο είναι σημαντικό, ενδιαφέρον επίσης, θεωρούμε εμείς, είναι να δούμε πώς χρησιμοποιείται το φύλλο αυτή τη στιγμή στη διαμόρφωση των τιμών στον ασφαλιστικό τομέα και πώς θα επηρεάσει η απόφαση αυτή τα ασφάλιστρα και άρα και τους πελάτες των ασφαλιστικών εταιριών. Όπως είπε και η Ευρωπαϊκή εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όλα τα κράτη-μέλη χρησιμοποίησαν την δυνατότητα της εξαίρεσης. Άρα η εξαίρεση ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή για τον κλάδο ζωής. Σε, για τα άλλα προϊόντα κάποιοι χρησιμοποίησαν την εξαίρεση, κάποιοι όχι. Αν δούμε τον ασφαλιστικό κλάδο αυτό καθεαυτό, είναι σημαντικό να σημειώσετε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες χρησιμοποιούν το φύλλο για τα προϊόντα τους μόνο αν το φύλλο επηρεάζει τα προϊόντα αυτά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιείται το φύλλο ως κριτήριο όταν κάνουμε ασφάλιση κάποιου κτηρίου. Αλλά για άλλα προϊόντα για την ασφάλεια ζωής. Παραδείγματος χάρη το φύλλο επηρεάζει επειδή είναι διαφορετικό το προσδόκιμο ζωής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη η μέση διαφορά είναι 6,5 χρόνια μεταξύ ανδρών και γυναικών. Χρησιμοποιείται επίσης και σε προϊόντα που σχετίζονται με την ε, υγεία Παραδείγματος Υπάρχουν βεβαίως ορισμ... υπάρχουν διαφορές. Υπάρχει ο καρκίνος του προστάτη και ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας που είναι εξαρτώνται από το φύλλο. Μοιραία λοιπόν τα προϊόντα που σχετίζονται με την υγεία επηρεάζονται από το φύλλο επίση υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία η ιατρική χρησιμοποιεί διαφορετικές θεραπείες για ορισμένες νόσους ανάλογα με το φύλλο και προφανώς οι διαφορετικές θεραπείες κοστίζουν διαφορετικά το ίδιο και για την ασφάλεια των αυτοκινήτων είτε μας αρέσει είτε όχι είναι σαφές ότι ιδιαίτερα για τους νέους οδηγούς κάτω των 25 ετών τα στατιστικά στοιχεία για ατυχημάτων, ατυχημάτων είναι διαφορετικά ανάλογα με το φύλλο και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη όταν διαμορφώνουμε τις τιμές για τέτοιου είδους προϊόντα. Το ίδιο συμβαίνει και τα δυστυχήματα για, τα, για άλλα ατυχήματα και εδώ οι στατιστικές μας δίνουν στοιχεία οι γυναίκες έχουν λιγότερα ατυχήματα και γι' αυτό, τουλάχιστον στο σπίτι και γι' αυτό α, χρησιμοποιείται το φύλλο και τα ασφάλιστρα για τις γυναίκες σε όλες αυτές τις κατηγορίες που σας ανέφερα είναι χαμηλότερα γιατί οι γυναίκες θεωρείται ότι έχουν ότι παρουσιάζουν χαμηλότερους κινδύνους Βάσει τώρα της ισότητας των φύλων και αν δεν ισχύει το 5-2 της οδηγίας, τότε θα πρέπει και εμείς να εξισώσουμε τα ασφάλιστρα, οπότε θα αυξηθούν τα ασφάλιστρα για τις γυναίκες. Και τώρα είχαμε στο κλάδο ζωής, σημαντικότερος κλάδος για το τομέα μας. Ένα προϊόν που παίζει τεράστιο ρόλο ο παραδείγματος χάρη στις μελλοντικέ επενδύσεις είναι η υποθήκη αυτό για να πάρετε υποθήκη είστε υποχρεωμένος να κάνετε ασφάλιση ζωής και εδώ οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Οπότε η ασφάλεια ζωής είναι φτηνότερη για τις γυναίκες. Αλλά εάν δεν χρησιμοποιήσουμε την εξαίρεση του 5-2 και χρησιμοποιήσουμε αυστηρά ίση μεταχείριση των δύο φύλων, τότε τα ασφάλιστα των γυναικών θα αυξηθούν. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα προϊόντα ε, τα οποία ίσως σας ενδιαφέρει να δείτε. Αν αγοράστε, παραδείγματος χάρη ε, annuity και ε, από εκεί και πέρα ε, κατά καταθέσετε ένα σημαντικό ποσό από το οποίο παίρνετε αμηνιές ε, δόσεις ε, τα, και εδώ ή τα ασφάλιστα για τις γυναίκες είναι φτηνό, το προϊόν είναι φτηνότερο για τις γυναίκες ε, γιατί το προσδόκιμο λόγι ζωής είναι μεγαλύτερο. Οπότε θα, η αύξηση των ασφαλίστρων εδώ θα ήταν ένα άλλο αρνητικό αποτέλεσμα και ενδεχομένως θα οδηγούμεθα σε μια κατάσταση κατά την οποία κάποιοι δεν Κάποιοι άνδρες ας πούμε δεν θα χρησιμοποιούσαν την ανιούητη μέσω ασφαλιστικών εταιριών αλλά θα πήγαιναν στις τράπεζες. Βεβαίως εκεί υπάρχουν άλλα προβλήματα. Και ε, αυτά θα πρέπει να συνυπολογιστούν βεβαίως. Εν πάση περιπτώσει σταματώ εδώ και είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας και θα ήθελα ε, με την αυτή τη στιγμή να ευχαριστήσω ένα καινούργια συνάδελφο. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας, καλώς ήρθατε στην, ε, ε, μας. Καλωσορίζω λοιπόν την κυρία Σακλέβα από την Σλοβενία. Και τώρα Προτείνω να συνεχίσουμε με τη συζήτησή μας και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Γκουρμάη που είναι η συγγήτριά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, χαίρομαι που συμμετέχω σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια και στην εργασία αυτή της Επιτροπής και βλέπουμε εδώ την ε, Γενική Γραμματέα της ε, Ευρωπαϊκής Συνδικαλιστικής Οργανώσεως Γυναικών και νομίζω ότι ε, θα μας βοηθήσει πολύ στον τομέα αυτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την βοήθειά της στην οργάνωση αυτής της παρουσίασης της Επιτροπής Γυναικών. Και βεβαίως λυπάμαι ότι η Σα δεν είναι εδώ, διότι καλό θα ήταν να μπορέσουμε να ε, συζητήσουμε το θέμα αυτό και να παρίστανται διότι ε, εάν υπάρχει τέτοιο σύστημα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ε, θα εξασφαλίζεται η ισότητα των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, στο ε, ισογγής μέλλον ελπίζω ότι βάσει αυτής της εργασίας ε, θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση των λαών της Ευρώπης ε, που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Συνοψίζω το τι έχει συμβεί μέχρι στιγμής, φαντάζομαι ότι γνωρίζετε. Ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απεφάνθη ότι το άρθρο 5 ήταν ενάντιο εις το Ευρωπαϊκό ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με την ισότητα των φύλων και την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και Και ε, το άρθρο 5 παράγραφο 2 ε, ε, προέβαινε σε διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών και το πιο προφανές παράδειγμα ήταν ε, αυτό των ε, φθηνών ε, ασφαλίσεων που καλύπτουν τα πιο συχνά ατυχήματα και ο νομοθέτης δεν έχει θέσει ένα χρονικό περιθώριο για την επανόρθωση και απλώς απεφανθεί ότι δεν μπορεί να συνεχίσει στο δυναικές μια τέτοια κατάσταση και ε, θεώρησε ότι καθίσταται ανίσχυρο από τις 21 Δεκεμβρίου του 2012 και ενημερώνει τους παρόχους υπηρεσιών. Διαφή είναι δηλαδή επαρκή χρόνο για να γίνουν οι αλλαγές. Πρέπει να ολοκληρωθεί η έκθεση, η έκθεση ε, της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά τώρα δεν είναι κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε τις αλλαγές. Απλώς αποδεικνύεται ότι ε, θεωρείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι υπάρχει ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, αλλά μπορεί ο ασφαλιστικός τομέας να προσπαθήσει να αυξήσει τις τιμές ε, γιατί ε, ίσως ε, θεωρούν ότι θα τους είναι πιο δύσκολο να καλύψουν τον κίνδυνο. Υπάρχει μια οικονομική κρίση άρα σε αυτό το κλίμα δεν θα είναι εύκολο να εφαρμοστεί το, αυτή η απόφαση και θα επανέλθω στο στοιχείο αυτό αργότερα. Τρίτον, σε λίγους μήνες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αρχίσει να αξιολογεί την εφαρμογή της ε, ε, διακρίσει ε, της οδηγίας του Συμβουλίου 2004 κάθετος 113 αλλά δεν θα, μας, δεν θα θεωρήσουμε ότι έχουμε αποτύχει απλώς για την δικαστική απόφαση της Τέστασα Απλώς θέλω να σας επισημάνω ότι όλη αυτή η διαδικασία δεν θα είναι απλή σε αυτό το πλαίσιο και ελπίζουμε θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την εργασία μας γιατί ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει καθυστερήσει ε, την αξιολόγηση πρώτον λόγω της εκδόσεως της απόφασης για την τέστασα και ε, ε, τώρα μας έχει ε, παρουσιάσει μία πλήρη απόφαση, αλλά θα πρέπει να ολοκληρώσει και την αξιολόγησή της για να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά. Είναι βασικό δηλαδή να υπάρξει σωστός προγραμματισμός και αναφέρατε τις δύο βασικές ημερομηνίες ορόσημα του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να εξασφαλίσω ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών ε, στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και θα προτιμούσα μία ε, επιχείρηση να βρει έναν καλύτερο τρόπο να μην αυξήσει τις τιμές γιατί μπορεί να χάσει τους πελάτες της και δεν θέλω οι πελάτες να χρειαστεί να πληρώσουν περισσότερα για για να μην υπάρχουν διακρίσεις. Θα ήθελα λοιπόν την αξιολόγησή σας, θα ήθελα όμως να σας πω ότι αν έπρεπε να επιλέξω για το ποιον θα έπρεπε να προασπίσω, θα προάσπιζα τον καταναλωτή χωρίς να το ξανασκεφτώ και βεβαίως αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ε, ο τομέας των ασφαλιών. Ξέρω ε, τις ε, ανάγκες που υπάρχουν για την κεφαλαϊκή επάρκεια σύμφωνα με το Solvency 2 και ε, ο στόχος μου ε, δεν είναι ε, να επιβάλλω μια απόφαση. Είμαι ανοιχτή σε όλους τους συμβιβασμούς, αλλά νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι θα ήταν άδικο να πληρώσει κανείς υψηλότερο τίμημα για να αποφύγει διακρίσεις. Δεν είναι αυτός ο στόχος της προσπαθίας μας. Ε, επίσης δεν υπάρχει αναδρομική εφαρμογή της απόφασης αυτής. Δεν χρειάζεται να σας πω την ε, αγωγή στην Ουγγαρία γιατί θα είχα προβλήματα και αναφέρεται οι ε, ε, συμβόλαια τα οποία υπεγράφησαν μετά τις 21 Δεκεμβρίου 2007. Αλλά πρέπει να δούμε πώς ε, θα συνδυαστούν οι αναθεωρήσεις των συμβολέων με τις νέες παροχές για να αποφύγουμε αμφισημίες. Ε, διότι πιστεύω ότι δημιουργούνται προβλήματα με τα ισχύοντα συμβόλαια και θα ήθελα να γνωρίζω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να τροποποιήσει την οδηγία σχετικά με αυτό το πρόβλημα κατά τρόπον ώστε να αξιολογήσουμε και αυτό το στοιχείο ο, κατά τη διάρκεια των εργασιών μας Επίσης ε, προτείνατε να συναντηθούμε με τους επικεφαλείς του κλάδου το Σεπτέμβριο. Μπορείτε παρακαλώ να μας δώσετε μία πιο πλήρη εικόνα για το τι θα προβλεφθεί σε αυτές τις συνεδριάσεις. Δεν θα επαρκέσει μία συνεδρίαση, θα χρειαστούν πολλές. Και δεν φτάνει να είναι ε, μόνο ο Επίτροπος ή ε, ε, ε, ε, αντικαταστάτριά της αλλά θα χρειαστεί να υπάρξουν πολλοί οι οποίοι θα συνεργαστούν και θα πρέπει η συνεργασία αυτή να διεξαστεί σωστά όταν θα έχουμε τα συμπεράσματα καλό θα ήταν να το γνωρίζουμε εγκαίρως και θα ήθελα να ξέρω εάν θα ε, δημοσιευθούν εγκαίρως. Ε, το ερώτημα είναι με πόση ειλικρίνεια και πόσο ανοιχτά θα γίνει αυτή η εργασία και το έβδομο μου σημείο είναι ότι ξέρω ότι ε, η ασφάλιση τώρα απαιτεί ε, να εφαρμόσει κανείς περισσότερο το άρθρο 5 παράγραφος 2 και ε, να δούμε ότι δεν υπάρχουν διακρίσεις και μέσω και για τη μεταχείριση των ε, ε, των ασφαλισμένων του ιδίου φύλου. Ποια είναι η γνώμη της Επιτροπής επ' αυτού. Και έρχομαι τώρα στο σημείο 8 και απευθύνομαι εις ε, τους συναδέλφους γιατί νομίζω ότι είναι κάτι που μας απασχολεί όλους. Θα χρειαστεί να συνδυάσουμε αυτό το πρόβλημα και σε άλλες διακρίσεις που υπάρχουν στο νομοθετικό πλαίσιο. Δηλαδή θα ήθελα να ζητήσω τους συναδέλφους αν έχουν ιδέες, να μου τις ε, μεταδώσουν ε, και θα τις ενσωματώσω με τα χαράς. Είναι ένα πολύ βασικό θέμα. Επιζητούμε να υπάρξει ίση μεταχείριση κατά προτεραιότητα, αλλά ε, χρειάζεται να έχει κανείς και να χρησιμοποιήσει και το καλό αλλά και το κακό από την άλλη πλευρά σαν τρόπο μεταχειρήσεως και ε, νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε όπως προχωρήσαμε στο θέμα της περιφοράς ε, της κινητής τηλεφορίας. Ευχαριστώ κυρία Γκουρμάη. Νομίζω ότι συμφωνούμε μαζί σας όταν λέμε ότι αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό και τώρα θα, να ξεκινήσει η συζήτηση και ίσως θα μπορούσα να δώσω το λόγο στον κύριο Ρωμέβα. Θα ήθελα να τονίσω πρώτα πρώτα το θέμα το οποίο συζητούμε έχει πολλές ε, και διαφορετικές ε, πλευρές ε, δεν είναι εύκολο να έχει κανείς μονοσήμαντη άποψη. Βεβαίως όλοι θέλουμε, ε, είμαστε εναντίον των διακρίσεων και όλοι θέλουμε να υπάρχει ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση σε υπηρεσίες και προϊόντα. Όμως υπάρχει και κάτι τι άλλο που πρέπει να σημειώσουμε για την ε, Είμαι εισηγητής για την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών όσον αφορά την ίση μεταχείριση και τη μη διάκριση λόγω θρησκευτικών πεπιθήσεων, εκτός δουλειάς, ε, λόγω ε, θρησκευτικών πεπιθήσεων και τα λοιπά. Και βλέπουμε, βλέπω ότι πραγματικά εδώ στο θέμα αυτό γίνονται προσπάθειες και από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όλοι οι άλλοι ενδιαφερόμενοι. Όμως τα πράγματα είναι ιδιαίτερα περίπλοκα εκεί και οι παράμετροι που πρέπει να λάβουμε υπόψη πάρα πολλές. Εδώ τα πράγματα είναι πιο απλά γιατί έχουμε την απόφαση του, του ΔΕΚ. Ε, Μιλάμε για ασφαλιστικές εταιρείε βεβαίως, ένα πολύ συγκεκριμένο κλάδο και δεν μιλάμε μοναχά για φύλλο, μιλάμε για ηλικία. Άλλη μια παράμετρος πρέπει να ληφθεί υπόψη και εδώ. Και βεβαίως καταλαβαίνω την ανάλυση που έκαναν ορισμένοι και που είπαν ότι προφανώς ιδιαίτερα λόγω της οικονομικής κρίσης την οποία βιώνουμε ε, είναι ε, σημαντικό να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλές και να μην ε, οδηγηθούμε σε ψηλότερα, σε ακριβότερα προϊόντα λόγω της μη διάκρισης. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν πρέπει να υπονομεύσουμε την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Δεν θεωρώ ότι η οικονομική προσέγγιση είναι σωστή. Εγώ διαφωνώ λοιπόν για το ότι πρέπει να, να βασιστούμε σε οικονομικά επιχειρήματα. Ως εισηγητής για παρόμοια θέματα αλλά ε, σας είπα για θέματα ε, εκτός δουλειάς και ε, για θρησκευτικέ πεπιθήσεις και τα λοιπά. Δεν αρκούν τα στατιστικά στοιχεία. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να βασιστούμε στα στατιστικά και οικονομικά στοιχεία για να πάρουμε θέση εδώ. Θα πρέπει να προσεγγίσουμε το θέμα από ένα άλλο πρίσμα πιο ανθρώπινο, πιο α, θεωρητικό ενδεχομένως και βεβαίως υπάρχει η απόφαση που μας δίνει κάποιες ιδέες για το τι θα γίνει στο μέλλον γιατί εγώ πιστεύω ότι στο μέλλον θα έχουμε ίσως να εξετάσουμε και πάρα πολλές άλλες οδηγίες οι οποίες ε, άπτονται της ίσης μεταχείρισης ε, λόγω φίλου. Λοιπόν, μην κολλάμε στα στατιστικά και στα οικονομικά επιχειρήματα. Βεβαίως λύση δεν έχω να προτείνω, γενική λύση δεν έχω να προτείνω. Νομίζω ότι τις λύσεις θα πρέπει να τις βρούμε κατά περίπτωση και θεωρώ πω ότι είναι πολύ καλό το γεγονός ότι έχουμε στη διάθεσή μας την απόφαση του δικαστηρίου. Εύχομαι καλή επιτυχία στην εισηγήτρια και ελπίζω στο τέλος να καταλήξουμε σε μια συνενετική άποψη η οποία θα έχει σαν κύριο στόχο το να καταπολεμά τις ε, διακρίσεις. Ευχαριστώ κυρία Γιάννα έχει το λόγο τώρα. Shows I haven't been here long enough. Φαίνεται είμαι καινούρια και δεν τα έχω μάθει ακόμα. Λοιπόν, αυτή είναι από τις χαρακτηριστικές δύσκολες περιπτώσεις που κανείς δεν θέλει να την αναλάβει. Λοιπόν, εδώ η αποτίμηση του κινδύνου βασίζεται σε ορισμένα κριτήρια μεταξύ των οποίων και το φύλλο. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε και θα ήταν άδικο προς τις γυναίκες να το αγνοήσουμε. Ξέρω ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα των οδηγών γυναικών, ας πούμε. Βέβαια, όλα τα θέματα τα αφορά το φίλο, αλλά αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Δεν ξέρω ούτε εγώ τι ακριβώς να σας πω, ούτε τι θέλουμε, ποιος είναι ο στόχος μας περιμένω την υπόλοιπη συζήτηση. Καμιά φορά το θέμα της ισότητας ή ο αγώνας για την ισότητα μπορεί να καταλήξει σε ανισότητα, μεγαλύτερη ανισότητα. Έχω κάνει ορισμένε σημειώσει και λέω εδώ ότι οι γυναίκες μπορεί να είναι καλύτερες σε ορισμένους τομείς όπως στην οδήγηση. Αυτό δείχνει τουλάχιστον η υποτίμηση των κινδύνων από τους ασφαλιστές και όταν έγινε μια προσπάθεια να εξισωθούν οι κίνδυνοι με τον ανδρών ε, σημειώθηκαν μεγαλύτερα ατυχήματα. Κάντε μια προσπάθεια οι άντρες να μας φτάσετε κάποτε. Πρέπει όμως η αποτίμηση να γίνεται σωστά. Τώρα για την άνηση μεταχείριση, όντως δεν θέλουμε άνηση μεταχείριση, αλλά δεν θεωρώ τις ασφαλίσεις και τα κριτήρια που εφαρμόζουν ως ότι βασίζονται σε άνηση μεταχείριση το θέμα είναι οι πιθανότητες και οι κίνδυνοι. Έτσι το βλέπουν οι ασφαλιστές, όχι με αρχές. Το να ανήκει κανείς στο α ή το β γένος μπορεί να θεωρείται ως κάτι πιο επικίνδυνο από ότι να ανήκει στο άλλο. Δεν είναι θέμα ούτε ισότητα ούτε θεωρητικά φίλων. Έχετε όμως δίκιο, πρέπει να τα δούμε ατομικά και οι ασφαλίσεις αυτό κάνουν. Λένε ποιος είναι ο πιθανός κίνδυνος που αντιπροσωπεύει το τάδε άτομο για, το δίνα, για τη δίνα δραστηριότητα. Αν μια γυναίκα προκαλέσει τον ίδιο αριθμό ατυχημάτων με έναν άντρα θα εξισωθεί από τις ασφαλίσεις με τον άντρα. Και αυτά που θα πρέπει να πληρώνει θα είναι τα ίδια έχουν μεν έναν γενικό κανόνα αλλά τον προσαρμόζουν κάθε φορά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γι' αυτό δεν έχω καθαρές απόψεις, ε, πρέπει να δω τι άλλο θα μας πει η συγγήτρια και τι θα διαπιστώσει. Ευχαριστούμε κυρία Γιάννα Κουδάκη. Κυρία Κώστα. Μια Ιταλική εφημερίδα έγραψε τον τίτλο «Το παράδοξον της ισότητας», το οξύμορο της ισότητας. Δεν ξέρω τι σημαίνει ακριβώς. Α, φαντάζομαι ότι αυτά που θα πω μπορεί να μην είναι πολύ πολιτικός ορθά, αλλά τι έγραφε, ότι υπάρχει στην πράξη άνηση μεταχείριση κατά των ανδρών, νομικά και πολιτικά όμως, όπως το είπε και η συγγήτρια και συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Νομικά και πολιτικά λοιπόν η απόφαση βασίζεται στη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων για να ακυρώσει το σχετικό άρθρο της οδηγίας και λέει ότι πρόκειται για άνηση μεταχείριση ενώ οι κίνδυνοι αποτιμούνται με καθαρά στατιστικό τρόπο και όχι ατομικό. Αυτό είναι το παράδοξο και το οξύμορο. Εμείς είμαστε πολιτικοί και πολιτικές και επομένως πρέπει να δούμε τι επιπτώσεις μπορεί να έχει η άνηση μεταχείριση με βάση το φύλλο στις ασφαλίσεις. Και εγώ δεν θα ήθελα να αυξηθούν τα πριμ και να δημιουργείται άνηση μεταχείριση, αλλά διάβασα προσεκτικά την απόφαση και είδα ότι ό,τι αφορά την πρόσθετη προστασία για τη μητρότητα, ας πούμε, δεν καλύπτεται. Για τις ασφάλειες ζωής, ε, αυτοκινήτων, ε, για ατυχήματα κλπ, οικιακά ατυχήματα, για όλα αυτά μόνο στα οικιακά τυχήματα σημειώνονται περισσότερες περιπτώσεις για γυναίκες και άρα μόνο εκεί μπορεί κανείς να πει ότι ωφελούνται οι άντρες. Πιστεύω και εγώ ότι η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σε επίπεδο αρχών είναι μεγάλη αλλά πρέπει να καταλάβουμε καλά τι θα γίνει αν η εφαρμογή δεν είναι επαρκώς δικαιολογημένη. Μπορεί να έχει τεράστιες επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Και η κυρία εισηγήτρια και άλλοι είπαν ότι πρέπει να υπάρχει απόλυτη νομική βεβαιότηση. Καταρχήν, ως προς την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει να εφαρμόζεται το νέο καθεστώς. Δεύτερον, τα εθνικά συστήματα όλα επέλεξαν να εφαρμόσουν τις εξαιρέσεις. Δηλαδή, να τα ξαναδούν όλα από την αρχή. Οι χώρες που επέλεξαν την οδηγία, ίσως από αδράνεια,

που από το 12 προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή. Η καθυστέρηση αυτή είναι ακόμη ένα εμπόδιο. Γιατί επειδή υπάρχει καθυστέρηση δεν εκλήθησαν τα κράτη-μέλη και οι ασφαλιστικές εταιρείες να αλλάξουν μέθοδο. Γενικά σημειώνεται λοιπόν μια καθυστέρηση εδώ για την οδηγία και η απόφαση του δικαστηρίου λέει απλώς ότι δεν μπορεί μετά το 12 να συνεχίσει να εφαρμόζεται η εξαίρεση. Ενώ μέχρι τώρα η οδηγία έλεγε ότι πρέπει να γίνει μελέτη αξιολόγησης μετά από τρία χρόνια και αν διαπίστωνε τότε η Κομισιόν ότι το υπάρχον σύστημα με τα στατιστικά στοιχεία ήταν βιώσιμο, διαφανές και ενημερωμένο, τότε μπορεί να χορηγούσε και νέα εξαίρεση. Ενώ η απόφαση λέει ότι μετά το 12 αυτό δεν γίνεται, αποκλείεται. Αυτή είναι η διαφορά. Πρέπει λοιπόν να έχουμε περισσότερα στοιχεία στην έκθεσή μας και περισσότερες και σαφέστερες πληροφορίες. Αλλά και εναλλακτικά σενάρια για να δούμε πώς θα μπορούσαμε και εμείς να επιλέξουμε. Ούτως ή άλλως θα χρειαστεί να αλλάξει το σύστημα. Αυτό είναι σαφές και ε, μοιάζει λιγάκι με τη συζήτηση για τις τράπεζες. Μπορεί να υπάρχει άνηση μεταχείριση με βάση την ηλικία όπως είπαμε για τις τράπεζες και εδώ. Για τα δάνεια μέχρι τώρα βασιζόμασταν στο κριτήριο της ιδιοκτησίας για υποθήκες ως εγγύηση. Σε περίπτωση όμως που δεν έχει κανείς τέτοια εγγύηση, οι τράπεζες κάνουν εξαιρέσεις, δηλαδή μια ειδική μελέτη εξατομικευμένη για τον κίνδυνο που μπορεί να εκπροσωπεί να εκπροσωπεί. Η Κομισιόν έθεσε το ερώτημα αυτό και νομίζω ότι και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να το θέσει γιατί μπορεί να υπάρχει τεράστια επίπτωση αν δεν λάβουμε υπόψη κανένα μέτρο. Ευχαριστούμε κύριε Κώστα. Κυρία Σεσίλ Κρανοβάλ. Ευχαριστώ πολύ. Το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών εκπροσωπεί πολλές γυναικείες οργανώσεις στην Ευρώπη, πάνω από 2.000 και ε, εμείς χαιρόμαστε για τη συζήτηση αυτή γιατί θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι όταν εγκρίθηκε η οδηγία είχαμε ταχθεί κατά της εξαίρεσης και αυτό είχε πει τότε και η Κομισιόν και η Επιτροπή σας. το θέμα αυτό πάντοτε το συνδέαμε με το ευρύτερο θέμα των συντάξεων των γυναικών και των διαφορών μεταξύ των συντάξεων των φύλων. Μιλάμε για τα δημόσια συστήματα συνταξιοδότησης που είναι τόσο ανεπαρκή που αναγκαζόμαστε να κάνουμε και συμπληρωματική ασφάλιση ιδιωτική. Επειδή λοιπόν αναγκαζόμαστε να απευθυνθούμε και στα ιδιωτικά συστήματα συνταξιοδότησης, θεωρούμε ότι τέτοιου είδους εξαιρέσεις αν επιτραπούν, αν συνεχίσουν να επιτρέπονται, θα μειώσουν ακόμη περισσότερο τα έσοδα των γυναικών στη σύνταξή τους. Γιατί οι γυναίκες ήδη έχουν χειρότερες συνθήκες και αυτά όλα πρέπει να πάψουν. Γι' αυτόν τον λόγο είμαστε υπέρ της αλλαγής του συστήματος. Όσο για το κόστος που θα επιφέρει η αλλαγή, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί να αυξηθεί. Αντίθετα πρέπει να γίνει μια ανακατανομή του κόστους και αυτά που λέμε τα λένε και οι οργανώσεις των καταναλωτών ότι δηλαδή τα κριτήρια που δεν μπορεί να ελέγξει ένα άτομο όπως το η φυλή δεν μπορεί να λαμβάνονται υπόψη ενώ κριτήρια τρόπου ζωής θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αλλά ούτε το φύλλο ούτε η φυλή. Επίσης, σε πολλές χώρες βασίζονται σε πριμ με βάση προηγούμενα στατιστικά στοιχεία για ατυχήματα. Αν φανεί ότι οι γυναίκες οδηγούν καλύτερα, αυτό σημαίνει απλώς ότι γενικά οι καλύτεροι οδηγοί θα πληρώνουν λιγότερο, όχι ειδικά οι γυναίκες. Ελπίζουμε λοιπόν να καταλήξουν όλα αυτά θετικά για τις γυναίκες ως πελάτησες των ασφαλιών για να σταματήσει πια αυτή η εξαίρεση που τη θεωρούμε ως μη συνεπή με τους στόχους της οδηγίας. Ευχαριστώ πολύ και τώρα θα επανέλθω στην κυρία Κόλλερ εκ μέρους του κλάδο των ασφαλιστών. Ναι, θα ήθελα να κάνω μερικά σχόλια. Αρχίζω λέγοντας ότι όταν ότι αν δούμε πώς διαμορφώνονται οι τιμές των ασφαλίστρων και τα λοιπά, δεν υπάρχει πραγματικά διάκριση ανάλογα με το φύλλο. Αλλά υπάρχουν διαφορές επί τη βάση άλλων κριτηρίων και επί τη βάση της αποτίμησης του κινδύνου. Η αποτίμηση κινδύνου βασίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία διαχρονικά, ας πούμε. Η το σίγουρα η παράμετρος του φύλου δεν είναι η μόνη παράμετρος που χρησιμοποιείται για να αποτιμηθεί ο κίνδυνος και άρα ε, να οριστούν οι τιμές. Και αυτό μπορούμε να το καταδείξουμε με στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν. Εκείνο που κάνουμε είναι να βλέπουμε κατά περίπτωση τα πράγματα και παρόμοιες περίπτωσεις πτώσεις τις αντιμετωπίζουμε με παρόμοιο τρόπο. Αυτό που είπε η εκπρόσωπος από το λόμπι των γυναικών που είπε ότι τελικά δεν πρέπει να υπάρχει διάκριση και στο τέλος πρέπει να γίνει ανακατανομή του κόστους αυτό είναι μια απλοϊκή προσέγγιση είμαι αποχρεωμένη να πω εντάξει, συμμετοχή ε, στα δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα είναι γενική και όλοι τις ίδιες εισφορές και πληρώνουν το ίδιο. Αλλά όταν είμαστε στον ιδιωτικό τομέα, ιδιαίτερα εμείς στις ασφαλιστικές εταιρείες, ε, ε, ε έχουμε κάποιες υποχρεώσεις για να μπορούμε να καλύψουμε συγκεκριμένους κινδύνους και οι κίνδυνοι αυτοί πώς να το κάνουμε πρέπει να το παραδεχθούμε είναι διαφορετική για τις γυναίκες εν πάση περιπτώσει δεν μπαίνω σε άλλες λεπτομέρειες αλλά νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε ε, πώς αποτιμούμε τα πράγματα στον τομέα. Κυρία Τομπόη. Yes, madam. Just... Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα πρακτικής εφαρμογής και όλα αυτά που αναφέρθηκαν εδώ για ε, έμεση αν θέλετε διάκριση έμεσες διακρίσεις και τα Ξέρουμε τα επιχειρήματα και των κρατών μελών και των ασφαλιστικών εταιριών και τα Είναι πολύ ε, σημαντικά όλα αυτά. Γι' αυτό θέλουμε να γίνουν συζητήσεις σε, από όλους με όλους τους ενδιαφερόμενους. Εμείς ελπίζουμε ότι στη συνάντηση θα οργανώσουμε το φθινόπωρο και από τις απαντήσεις που θα, ναι, θα απαντηθούν πολλά ερωτήματα και έχουμε και ένα ερωτηματολόγιο το οποίο στείλαμε εν ώψη της συνάντηση αυτής το οποίο ελπίζουμε θα μας δώσει σημαντικές απαντήσεις και αυτό. Ευχαριστώ. Και τώρα δίνω το λόγο στο, στην εισηγήτριά μας την κυρία Γκουρμάη. Καταρχήν θέλω και πάλι να ευχαριστήσω όσους συμμετείχαν στη συζήτηση και ελπίζω ότι είναι καλό να γνωρίζει κανείς τις διάφορες πτυχές όπως άλλωστε και τις διάφορες απόψεις επί του θέματος αυτού. Και ε, επειδή είναι η περίοδος της Ουγγρικής Προεδρίας, πολύ θα με ενδιαφέρει να ακούσω και τη θέση της ε, ε, Προεδρίας του Συμβουλίου αυτή την εποχή. Ευχαριστώ όλους για, τις, για τα σημαντικά σχόλια. Όπως είπα από την αρχή δεν πρόκειται να είναι κάτι το εύκολο και ελπίζουμε όσοι πρεσβεύουν την ε, πρόθεση ίσης μεταχείρισης ότι θα υπάρξει μια σωστή λύση και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζουμε ότι θα διαχειριστούμε σωστά το θέμα αυτό αλλά θα πρέπει να συνεργαστούμε στενά καθ' όλη τη διαδικασία να ξέρουμε τι σκέφτονται οι ε, ασφαλιστικές εταιρείες και να καταλήξουμε ε, σε ένα καλό συμβιβασμό. Σας ευχαριστώ και χαίρομαι ιδιαιτέρως που ήρθε η Σεσίλ γιατί και αυτό είναι βασικό να συμμετέχουν και οι περιβαλλοντολογικές οργανώσεις. Ευχαριστώ κυρία Γκουρμάη και νομίζω ότι αυτό ολοκληρώνει το θέμα αυτό και θα επανέλθουμε. Τώρα το επόμενο είναι το 4 και εδώ είναι η πρόταση ε, εκθέσεως σχετικά με την κατάσταση των γυναικών που πλησιάζουν τη ηλικία συνταξιοδότηση Η συγγήτριά μας επ' αυτού για την Επιτροπή είναι η κυρία Μπάουερ και η έκθεση θα εξετάσει μία διπλή ε, διάκριση εναντίον των γυναικών είτε για κοινωνικά θέματα είτε για θέματα αγοράς εργασίας οπότε ε, αναφέρεται σε δύο σημεία δηλαδή και στο φύλλο και στην ηλικία ε, και εξαρτάται ε, από αυτό η τύχη των γυναικών μεγαλύτερης ηλικίας και θα ακούσουμε με τα προσοχή ό,τι έχει να μας πει η συγγήτρια. Επιπλέον η συγγήτρια ε, δεν εξετάζει μόνο την απασχόληση των γυναικών πέραν των 50 ετών, αλλά και την ε, κατάσταση των ε, γυναικών που αναλαμβάνουν ε, έργο περίθαλψης και ε, θα τονιστεί και αυτό το θέμα. Η συγγήτρια θα παρουσιάσει τώρα την πρότασή της και έτσι χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση δίνω το λόγο στην κυρία Μπάουερ ε, για να μας το παρουσιάσει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι εδώ μιλάμε για γυναίκες πέραν των 50 ετών. Καμιά φορά ενδέχεται να βρείτε στο κείμενο και άλλη ταξινόμηση ηλικίας διότι ε, δεν υπάρχουν πλήρεις και αξιόπιστες στατιστικές για τις ηλικιωμένες γυναίκες και αν γίνει ε, μία ε, κατανομή κατά ηλικία μεταξύ των φίλων βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορές. Άλλοι μιλάνε για 45-55, άλλοι μιλάνε για 50 έως 60 ετών. Προσπαθούμε λοιπόν να ε, εστιαστούμε στις γυναίκες οι οποίες είναι πέραν των 50 ετών. Θα ήθελα αν έχετε χρόνο να μπείτε στο Google και ε, να κοιτάξετε στατιστικά ε, στοιχεία για αυτή την περίοδο ηλικίας και βλέπετε πάρα πολλά στατιστικά στοιχεία Άρα ε, όντως υπήρχε ανάγκη για την έκθεση αυτή ε, και καλό είναι να ζητήσουμε πιο ασφαλείς ε, στατιστικές και νομίζω ότι αυτή η περίοδος είναι αποφασιστική διότι από την κατάρτιση της στρατηγικής το 2020 όπου υπάρχει στόχος απασχόλησης 55 100 των ανδρών και γυναικών βλέπουμε ότι οι γυναίκες πέραν των 55 μέχρι 64 ετών απασχολούνται μόνον κατά 37%. Και όσον αφορά το θέμα της ίσης μεταχείρισης βλέπετε ότι κάτω των 30 ετών απασχολούνται μόνο 8% των γυναικών και από 50 έως 59% η διαφορά είναι 22,5% στην απασχόληση. Ένα ακόμη στατιστικό στοιχείο, 58% των Ευρωπαίων όχι μόνο σε αυτήν ε, την ε, ηλικία, αλλά σε όλα τα ευρωπαϊκά στοιχεία ε, αποδεικνύουν ότι υπάρχει σημαντική διάκριση σχετικά με την ηλικία και οι γυναίκες θεωρώντουσαν ότι γερνάνε πολύ πιο νωρίς, πολύ πιο νωρίς από τους άντρες. Οπότε, εάν δουλεύετε σκληρά θα δείτε ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικά αποτελέσματα σχετικά με αυτό το θέμα της ηλικία σε πολλά σημεία. Προσπάθησα λοιπόν να διαπιστώσω τι συμβαίνει. Οι γυναίκες προχωρούν στην ε, πρόορη συνταξιοδότηση πολύ πιο γρήγορα. Καταρχήν, διότι υπάρχει μία σαφής διάκριση στην αγορά εργασίας. Ε, could you, Και βλέπετε να υπάρχει μία διάκριση και στους μισθούς και κάποια ποίηση για να φροντίσουν τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας. Δηλαδή εγώ όταν εγώ ο, και ξεκίνησα αυτή τη ε, διαδικασία είδα ότι ουσιαστικά υπήρχε ή ε, ε, κάποια διάκριση στη δεκαετία των 30 ετών και των 40 ετών αλλά τώρα βλέπουμε ότι ουσιαστικά η μεγαλύτερη διάκριση είναι ε, στην ηλικία μετά των 50 ή ασχολείται ε, με ε, ε, τον ε, επαγγελματικό τομέα είτε όχι. Λοιπόν, καλό θα ήταν εις τον τομέα αυτό να γίνουν περισσότερες έρευνες διότι βλέπουμε ότι όσον αφορά τις έρευνες για την υγειονομική ασφάλεια των ε, γυναικών ε, παρουσιάζουν επίσης ε, κάποια διάκριση σε σχέση με τους άντρες. Απλούστατα θα έπρεπε να δούμε ε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις γυναίκες αυτές όταν πρέπει να υπάρξει περίθαλψή τους, διότι υπάρχουν ορισμένοι οργανισμοί πιο ανθρώπινοι και Μία καλή πρακτική ε, σε αυτό το τομέα ε, για το Λουξεμβούργο όπου ασφαλίζονται οι γυναίκες οι οποίες μένουν στο σπίτι τους ε, βάσει νόμου και περιθάλτονται κρατική δαπάνη. Και αυτό που είναι επίσης ενδιαφέρον είναι το παράδειγμα της Ουγγαρίας όπου οι παππούδες και οι γιαγιάδες έχουν δικαίωμα γονικής αδείας και Χρειάζονται περισσότερα τέτοια παραδείγματα βελτίστων πρακτικών και αυτό το οποίο θα ήθελα να αναφέρω επιπλέον είναι ότι ε, τα άτομα αυτά που ασχολούνται με την περίθαλψη ε, χρειάζονται και συμβουλή αλλά και άδεια ε, γιατί το τα καθήκοντα αυτού του, σε αυτό το τομέα θα αυξηθούν πολύ. Θα ήθελα λοιπόν να μας απασχολήσει περισσότερο η ε, προληπτική υγιεινή, ε, να υπάρξει καλύτερη παρακολούθηση ώστε να παραμείνουν πιο ενεργοί ε, πιο ενεργά τα άτομα σε αυτή την ηλικία και αυτό που μπορώ να πω σχετικά με τη γενιά αυτή όσον αφορά την αγορά εργασίας, την ασφάλιση, τις συντάξεις, την ε, ε, φτώχεια γιατί προφανώς είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει. Βλέπουμε ότι η γενιά αυτή ε, συγκεντρώνει προϋποθέσεις σύμφωνη με τις οποίες ε, θα αντιμετωπίσει οικονομικά προβλήματα στη συνέχεια. Γι' αυτό και ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι του χρόνου θα συζητήσουμε ε, το θέμα της ε, γυράνσεως ε, με ενεργή δραστηριότητα και πρέπει να μας απασχολήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μπάουαρ. Τώρα η κυρία Γκουρμά έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πιστεύω πως το θέμα αυτής της έκθεσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και αποφασιστική σημασία για τις γυναίκες όπως συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν προκλήσεις οι γυναίκες ζουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το προσδόκιμο ζωής είναι μεγαλύτερο για τις γυναίκες από εκεί και πέρα έχουμε την στρατηγική της Λισαβόνας που δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες να συμμετάσχουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην ε, αγορά, να παραμείνουν ενεργέ στην αγορά εργασίας και όντως εν... Αλλά όμως παρόλα αυτά βλέπουμε ότι από μια ηλικία και πάνω 76,2% ε, των ατόμων στην αγορά εργασίας είναι άνδρες και το ποσοστό των γυναικών είναι πολύ χαμηλότερο. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέξουμε κάποιες ηλικίε όσον αφορά τις γυναίκες και για το κατά πόσο είναι πραγματικά ίση η μεταχείρισή τους ε, αυτή τη στιγμή. Από την άλλη μεριά η φτώχεια, η ένδυα, έχει και ένα ανθρώπινο πρόσωπο το οποίο δεν κοιτάζει φύλλα αυτή τη στιγμή ε, φτιάχνεται μια έκθεση για τις ε, συντάξεις και που είναι και αυτή σημαντική για τις γυναίκες που είναι κοντά στην ηλικία συνταξιοδότης ή, ή παίρνουν ήδη σύνταξη. Το μετά από την ε, διυπουργική του έψο ε, φτιάχτηκε το πρώτο κείμενο πρόχειρο αυτής της έκθεσης και κάπου με σοκάρισαν τα στοιχεία που περιλαμβάνει. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ε, ότι υπάρχουν προβλήματα και η έκθεση της Ρωμάνα Πλάμπ είδα που αναφέρεται στην ένδυα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είχε πραγματικά σοκαριστικά στοιχεία για το το ποσοστό των γυναικών μεταξύ των φτωχών της Ευρώπης που είναι πάρα πολύ ψηλό και βεβαίως όταν λέμε φτώχεια μιλάμε και για προβλήματα υγείας που απορρέουν από αυτήν και τα λοιπά. Αναφέρθηκε το πολύ καλό παράδειγμα της Ουγγαρίας στην οποία προβλέπεται ή κάποια άδεια για τους παππούδες και τις γιαγιάδες αντίστοιχη με τη γονική ε, άδεια. Αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ καλό παράδειγμα και βοηθά ε, στην όλη υπόθεση. Ε, κλείνοντας να πω ότι θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το αντικείμενο που συζητούμε αυτή τη στιγμή και για το οποίο είναι η συγγήτρια η Edith Bauer είμαι σίγουρη ότι θα φτιάξει μια πάρα πολύ καλή έκθεση και να πω και δύο λόγια γιατί ε, για το την ε, νεολαία και το πρόγραμμα νεολαίας 2020 και εκεί πρέπει να προσέξουμε την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών όπως κάνουμε όμως για τους νέους ε, και μιλάμε μια, μια ειδική έκθεση γι' αυτό με τον ίδιο τρόπο πρέπει να προβλέψουμε κάτι και για τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικία. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Γκουρμάη. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Λιωτάχ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω. Εδώ είμαι. Λοιπόν, ξαναρχίζω την αρχή και θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας την κυρία Μπάουερ για την παρέμβασή της και για τη δουλειά που κάνετε. Ε, να πω ότι συμφωνώ εμπολής με αυτά που είπε η κυρία Γκουρμάη. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το ε, ζήτημα που συζητούμε. Ε, ε, όπου δεν μιλάμε απλώς για διαφορές λόγω φύλου αλλά και για διαφορές λόγω ηλικίας. Είναι γεγονός ότι και βεβαίως ε, νομίζω ότι υπάρχει εδώ και ένας άλλος παράγοντας και ο πολιτιστικός παράγοντας ε, ενδεχομένως ε, διαφορετικές κουλτούρες υποχρεώνουν ε, τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας να κάνουν περισσότερα ή λιγότερα όσον αφορά τα μέλη της οικογένειάς τους ε, Πράγματι υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να εξετάσουμε και θεωρώ ότι αυτά που μας είπε η κυρία Μπάουερ είναι, ε, μας ε, πείθουν για το ότι θα φτιαχτεί μια πολύ καλή έκθεση στο τέλος. Ε, εγώ πήρα το λόγο για να τονίσω όμως και κάποιες άλλες πτυχές και κάποιες άλλες πτυχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Την σήμερον ημέρα άσχετα από, το, τις, από τις προσπάθειες που έχουν γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μη διάκριση μεταξύ των φύλων βλέπουμε να υπάρχουν να συνεχίζουν να υπάρχουν παραδοσιακοί ρόλοι στην κοινωνία μας ε, και μοιραία θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι γυναίκες αναλαμβάνουν περισσότερες ευθύνες και οι μεγαλύτερες ηλικία γυναίκες ακόμη περισσότερες δεν μπορούμε να γνω... αυτό θα πρέπει να τονιστεί στην έκθεσή σας κυρία Μπάουερ και Επίσης θα πρέπει να ε, συνειδητοποιήσουμε ότι το 2012 είναι το ευρωπαϊκό έτος για την ενεργή γύρανση όπως λέμε. Ναι, αλλά οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να μπορούν να είναι και ενεργοί. Θα πρέπει να έχουν το χρόνο να είναι και ενεργοί. Γιατί κάποιες γυναίκες πραγματικά αναλαμβάνουν πάρα πολλά σε μεγάλες ηλικίε που τις υποχρεώνουν να εγκαταλείψουν την ενεργή συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Εδώ χρειάζεται και μια αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών νομίζω εγώ. Αυτό θα πρέπει να το στην έκθεσή σας κυρία Μπάουερ θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τα Επίσης τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν κίνητρα για να συμμετάσχουν, να συνεχίσουν να παραμείνουν στην αγορά εργασίας οι γυναίκες. Πάρα πολύ ωραία. Ξέρω όμως πολλές γυναίκες μεγαλύτερης ηλικία που θα ήθελαν να μείνουν στην αγορά εργασίας αλλά δεν τους επιτρέπει ο, ο τρόπος ζωής τους ή η οικογένειά τους να κάνουν κάτι τέτοιο. Οι, οι γυναίκες προσφέρουν πολλά στην κοινωνία, όχι μόνο σαν μητέρα σε μικρότερη ηλικία, αλλά και όσον αφορά τη φροντίδα των ηλικιωμένων σε μεγαλύτερη ηλικία, τη φροντίδα των μικρών παιδιών, των εγγονιών, όπως αναφέρθηκε προηγούμενα. Προσφέρουν κοινωνικό έργο οι γυναίκες ε, ηλικία από τα 50 και πάνω και αυτό πρέπει να τονιστεί γιατί είναι και αυτό ενεργή συμμετοχή νομίζω άσχετα αν είναι ε, αν δεν βρίσκονται στην αγορά εργασίας αυτές οι γυναίκες επίσης κάτι τι άλλο θα ήθελα να τονίσω σχετικά με το, θέμα υγείας που αναφέρθηκε ε, πολλές φορές ε, μάλλον τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ε, να γίνονται ε, να υπάρχουν ερευνητικά προγράμματα για μ, όσον αφορά θέματα υγείας στα οποία η συμμετοχή των ανδρών ε, ή είναι μεγαλύτερη γιατί διότι ορισμένα συμπτώματα στις γυναίκες θεωρούνται απλώς συμπτώματα της μεγάλης ηλικίας και άρα αγνοείται ή, ή παραμελείται αν θέλετε ε, κάποια ομάδα ηλικιωμένων γυναικών. Αυτό θεωρώ ότι είναι ε, κακό. Επίσης ε, όσον αφορά τη φτώχεια γιατί ακούστηκε και αυτό η φτώχεια δημιουργεί προβλήματα υγείας. Η φτώχεια ε, η καταπολέμηση της φτώχειας θα έπρεπε να αφορά στον ίδιο βαθμό άνδρες και γυναίκες και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή γίνεται προσπάθεια να διασωθούν αν θέλετε οι νεότερες γυναίκες και οι άνδρες ασχέτως ηλικία. αυτό είναι διάκριση κατά των γυναικών μεγάλης ηλικίας η κυρία Κώστα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είναι μια δυνατότητα που θα μας δοθεί για να εμβαθύνουμε το θέμα αυτό διότι μέχρι στιγμής δεν έχει εξεταστεί επαρκώς. Πρώτη παρατήρηση. Είμαστε στην ε, πολύ ε, κοντά στην παραμονή του εορτασμού του έτους των σχέσεων μεταξύ των γενεών το 2012. Άρα μπορούμε ήδη να προετοιμάσουμε το έδαφος για τον εορτασμό αυτό. Και πολύ σωστά είπε η κυρία Μπάουερ ότι η ηλικία μεταξύ 50 και 60 ετών είναι πολύ ευάλωτη. Υπάρχουν πολλές ε, γυναίκες οι οποίες ε, ήδη αναχωρούν όχι ε, από ελεύθερη βούληση αλλά κατά ανάγκη σε πρόορη συνταξιοδότηση και έτσι τώρα θα μπορέσουμε να έχουμε μία ανάλυση των φαινομένων και των πρακτικών όπως άλλωστε και των λύσεων. Καταρχήν, η γονική άδεια είναι κάτι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν διάφορες λύσεις οι οποίες έχουν προταθεί στις διάφορες χώρες αλλά ε, πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν γυναίκες οι οποίες ε, είναι ε, αρχηγοί οικογενείας και είναι ευάλωτες. Ίσως υπάρχουν παιδιά που είναι ενήλικες νέοι αλλά σε μία ασαφή κατάσταση και άλλωστε τα χρόνια αυτά λαμβάνονται υπόψη και για τον υπολογισμό της συντάξεως. Άλλωστε στην Ιταλία υπάρχει ένα δικαίωμα για τις γυναίκες και όχι μόνον, το δικαίωμα δηλαδή να εργάζονται ε, ένα περιορισμένο ωράριο για να μην χρειαστεί να εξέλθουν από την αγορά εργασίας και το 80% των γυναικών στην Ιταλία έχουν χαμηλότερες συντάξεις από τους άντρες ιδίως διότι έχουν δυσκολία να παραμείνουν στην αγορά εργασίας και εδώ πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες χώρες όπου υπάρχει αυτό το οποίο ονομάζουμε σιωπηλέ σύνδρομες, ιδίως για γυναίκες οι οποίες ε, έχουν ε, συμβάλει ε, στην κοινωνική ασφάλιση αλλά όχι επαρκώς για να συνταξιοδοτηθούν διότι τα χρήματα αυτά πηγαίνουν σε ένα γενικό συνταξιοδοτικό ταμείο. Στην Ιταλία λοιπόν προσπαθούμε οι γυναίκες αυτές οι οποίες ε, έχουν ε, συμβάλει, ακόμη και αν το ποσό που έχουν καταβάλει δεν τους επιτρέπει να ε, συνταξιοδοτηθούν, να μπορέσουν να λάβουν πίσω το ποσό αυτό ή να ε, χαίρουν μίας μικτής κάλυψης. Δηλαδή οι γυναίκες που δεν έχουν το ελάχιστο, το, τις ελάχιστες προϋποθέσεις για να συνταξιοδοτηθούν θα έπρεπε ε, να ληφθούν υπόψη. Η κυρία Νίλσεν, ευχαριστώ. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω ε, την εισηγήτρια για την ενδιαφέρουσα αυτή έκθεση η οποία τονίζει την κατάσταση ε, ενός τμήματος του πληθυσμού το οποίο μας ενδιαφέρει είτε λίγο είτε δεν έχει εξεταστεί ε, σωστά και νομίζω ότι υπάρχουν και ε, λόγοι για τους οποίους πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Υπάρχει μία ειδική διάκριση που αναφέρεται ή στο φύλλο και είναι μία διάκριση η οποία συσσωρεύεται με άλλες, δηλαδή με αυτήν της ηλικία, αλλά και ειναι μια διακριση η οποια συσσωρευεται με αλλες δηλαδη με αυτή της ηλικια αλλα και της ε, σεξουαλικής προτιμήσεως, του χρώματος ε, του δέρματος ε, και οδηγεί σε πολλαπλές διακρίσεις συσσωρευτικά. Για να μπορέσει λοιπόν να διορθωθεί αυτή η συστηματική θα πρέπει να υπάρχει μία συμμετρική εφαρμογή των δημοσίων πολιτικών για να διορθωθούν οι επιπτώσεις ε, στην καριέρα, ε, στα διοδρομία ή στην επαγγελματική εξέλιξη και στην εργασία. Και θα πρέπει επίσης ε, να δουλέψουμε σκληρά μέσα στην κοινωνία για να μην υπάρξει πλέον τέτοιου είδους σχέσεις και ε, θα πρέπει να οργανωθεί ο χρόνος εργασίας των ανδρών και των γυναικών σε ζευγάρια όπου και οι δύο εργάζονται και αναφέρομαι στον κοινωνιολόγο Ντομινίκ Μεντά ο οποίος λέγει ότι οι ε, επιχειρήσεις παραμένουν ε, θέλουν να εθελοτυφλούν ε, ε, σχετικά με τις ανάγκες των εργαζομένων τους και θα έπρεπε να τους ανοίξουμε τα μάτια. Ε, αυτό θα ήθελα να πω κυρία Μπάουερ για να σας πω ότι συμφωνώ με την εργασία σας και ευχαρίστω θα σας στηρίξω. Ευχαριστώ και τώρα δίνω το λόγο στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στον εκπρόσωπο. Χαίρετε. Δεν είναι η κυρία Πέρεθ Γκουτμάγκετ, αλλά είμαι ο κύριος Μπαρμπόγια και σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει το βασικό αυτό θέμα και η οικονομική ανεξαρτησία είναι βασικό στοιχείο ε, για την εφαρμογή της στρατηγικής από το 2010-2015 διότι θεωρούμε ότι είναι ένα βασικό στοιχείο για να υπάρξει ίση μεταχείριση των ε, φύλων και παρόλο που δεν προβλέπεται το στοιχείο αυτό στη στρατηγική του 2020 δεν θα επιτύχουμε τον στόχο για τους άντρες και τις γυναίκες μεταξύ 20 και 65 ετών αν δεν καλύψουμε τα κενά στην ίση μεταχείριση και σε διάφορες άλλες βαθμίδες ηλικίας. Ε, θα βλέπουμε ότι υπάρχει ένα σχετισμό σε ορισμένε ηλικίε 70 με 75% και ε, από 55 μέχρι 64 υπάρχει ευρύτερη διάκριση και διαφορά. Οι γυναίκες απασχολούνται περίπου στο 38% ενώ οι άντρες απασχολούνται σχεδόν στο 55%. Και το... γι' αυτό και ξεκίνησε το πρώτο ευρωπαϊκό εξάμεινο με μία έρευνα ετήσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ίση μεταχείριση των φύλων διότι θεωρούμε ότι αυτό είναι βασικό για να εξετάσει κανείς ε, τι σχέση υπάρχει κατά τις ώρες εργασίας και μετά το σχολικό ωράριο διότι βλέπουμε ότι οι γυναίκες ε, ε, χωρίς να το επιθυμούν υποχρεώνονται να έχουν εργασία μερικής απασχόλησης και αυτό το πρόβλημα γίνεται πιο οξύ όσο γυράς και ο πληθυσμός. Οι γυναίκες ιδιαιτέρως έχουν μία ιδιάζουσα κατάσταση διότι πρέπει επίσης να στηρίξουν τα παιδιά να μεγαλώσουν μεγαλώσουν τα μέλη της οικογένειας και να φροντίσουν και τους γονείς και αυτό και στην αγορά εργασίες ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν τομές ε, και υπάρχουν ορισμένοι εργαζόμενοι που πρέπει να εγκαταλείψουν για να φροντίσουν τους γονείς τους. Ε, και εμποδίζεται κατά αυτόν τον τρόπο να υπάρξει μία φυσιολογική εξέλιξη στα διοδρομίες και μία παραγωγικότητα η οποία να βασίζεται στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων. Τέλος, ε, πρέπει να ε, αξιολογήσουμε όλα τα στοιχεία που μας δίδουν σχετικά με την ίση μεταχείριση των φύλων τα κράτη-μέλη. Διότι βλέπουμε ε, ότι στην αγορά εργασίας υπάρχουν διαταραχές και οι γυναίκες κινδυνεύουν από φτώχεια διότι ζουν περισσότερο χρόνο από τους άντρες και στα κράτη-μέλη βλέπουμε ότι ε, υπάρχει ε, ένα ποσοστό φτωχών γυναικών 20% έναντι 15% των ανδρών και θα πρέπει να αντισταθμίσουμε αυτή τη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας και να την στηρίξουμε με πολιτικές για την αγορά εργασίας διότι υπάρχει χαμηλό ποσοστό γονιμότητος επιμικίνεται η διάρκεια ζωής ε, και ε, η Ευρωπαϊκή Χρονιά, ο εορτασμός Ευρωπαϊκής Χρονιάς για την ενεργή γύραση θα μπορέσει να βοηθήσει την κοινωνία και να δείξει ότι υπάρχουν ευκαιρίες για τους άντρες και τις γυναίκες σε αυτή την ηλικία και ε, θα μπορέσει η πολιτική αυτή να ενταχθεί στις άλλες πολιτικές που αναφέρονται στη γύρανση διότι οι άντρες και οι γυναίκες εκτίθενται σε κινδύνους υγείας με διαφορετικό τρόπο και ακόμη και οι κοινωνικές υπηρεσίες που τους προσφέρονται επηρεάζονται από το φύλλο τους ε, διότι οι περισσότερες γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άνδρες αλλά όχι υποχρεωτικά σε καλή υγεία και πρέπει να λαμβάνει κανείς ε, υπόψη του κινδύνους οι οποίοι υπάρχουν σχετικά με την ε, υγεία και θα ε, συνεχίσουμε την εφαρμογή των πρακτικών, των βελτίστων πρακτικών προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων. Ευχαριστώ. Και δίνω τώρα το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Μπάουερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμφοβολή σας. Πρέπει να σας πω ότι προσπάθησα να σας δείξω ότι είναι απαραίτητο να εξετάζουμε την καριέρα των γυναικών σε όλη τους την ενεργό ζωή. και κάτι άλλο που τονίστηκε από τη συζήτηση είναι ότι υπάρχει το θέμα της συμφιλίωσης. Αν μιλήσουμε λοιπόν γι' αυτό, όταν μιλάμε γι' αυτό συνήθως εννοούμε μόνο τις νεαρές γυναίκες ή νεαρά ζεύγη με μικρά παιδιά. Η κατάσταση όμως αλλάζει τώρα, αλλάζει. μπορεί και πιο ηλικιωμένες γυναίκες. για τη συμφιλίωση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή. Γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τη φροντίδα ας πούμε των ε, εξαρτημένων ατόμων των μη ανεξάρτητων. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε πολλά, αλλά σε κάθε γνωμοδότηση, σε κάθε έκθεση υπάρχουν αυστηρά όρια στο μήκος τους. Παρακαλώ η γραμματεία να μου επιτρέψει να προσθέσω μια σελίδα λοιπόν. Αναμένω τροπολογίες, ναι. Φυσικά αντιμετώπισα τον πειρασμό να εξειδικεύσω το θέμα στην νεαρές ηλικίε, στη νέα γενιά, αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχει ο πειρασμός, αλλά πού θα σταματήσουμε στο κατέβασμα του ηλικία. Σε κάθε φάση της ζωής υπάρχουν προβλήματα και όλα συνδέονται. Προσπάθησα λοιπόν να θέσω κάποια όρια και να περιορίσω την προσοχή μου στο θέμα της ενεργού γυράνσεως. Τι εννοεί αυτό, τη δραστήριας γύρανση τι μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτές τις μεσόκοπες γυναίκες. Ευχαριστώ και αναμένω τις τροπολογίες σας. Ε, προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 31 Μαΐου και μετά το θέμα θα πάει με ορίζοντα για να πάει το θέμα στην Ολομέλεια ε, το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τώρα θα πάμε στην αίθουσα 3G2 του κτίριου ΑΣΠ για την κοινή αυτή συνεδρίαση με την Επιτροπή Ανάπτυξης που θα αρχίσει στις 11 η ώρα και θα ξαναγυρίσουμε στην αίθουσα αυτή το απόγευμα στις 3.